Madame le Président. Η Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Άρχεται η σημερινή συνεδρίαση. Να ξεκινήσουμε μία μικρή ανακοίνωση. Χθε αποφάσισε η συνέλευσή μας να προσθέσει στην ε, ημερήσια διάταξη για το μεσημέρι τις δηλώσεις του Συμβουλίου και τη Κομισιόν για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα την οικονομική κρίση. Θα ακολουθήσει γύρω των πολιτικών ομάδων ενημέρωσε το Συμβούλιο και η Κομισιόν ότι δεν θα είναι ε, παρόντες ε, στη συζήτηση αυτή. Μετά από επαφές που είχαμε όλες τις πολιτικές ομάδες, σας προτείνω ε, δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 2 του κανονισμού μας να τροποποιήσουμε αυτό το σημείο ως εξή. Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με θέμα την οικονομική κρίση. Θα ακολουθήσει γύρω των πολιτικών ομάδων. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την αλλαγή αυτής της μέρης για διάταξη. Αν όχι, εγκρίνεται η αλλαγή αυτή και περνάμε στις ε, προφορικές ερωτήσεις ε, προς ε, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2011 τα πρώτα διδάγματα. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Μπόλς ως συντάκτρα της ερώτησης. Δυόμιση λεπτά κυρία Μπόλς. Uh, um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια σημαντική καινοτομία στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς συγχρονίζονται οι μακροοικονομικές και οι φορολογικές διαστάσεις και ευθυγραμμίζονται οι στόχοι του 2020 στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Έχουμε επίσης τις εθνικές συστάσεις της ε, Κομισιόν που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο και έχουν στόχο να δώσουν μια κατεύθυνση εξ στα κράτη-μέλη όσον αφορά τους δημοσιονομικούς τους στόχους. Οι συστάσεις αυτές υιοθήθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούλιο μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν. Ως ε, μέρος του ρόλου του Κοινοβουλίου για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στο επίπεδο της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να συζητηθούν αυτές οι συστάσεις, αλλά και γενικότερα το αποτέλεσμα του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όλα αυτά τα ερωτήματα προς Κομισιόν και Συμβούλιο έχουν στόχο να αναθεωρήσουν το εξάμεινο για να βελτιωθεί. Συμβούλιο και Κομισιόν θεωρούν πως ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε το εξάμεινο και εάν δεν πήγαν όλα τέλεια, πώς θεωρούν πως θα πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία του χρόνου. Θεωρεί το Συμβούλιο πως οι αλλαγές που έγιναν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήταν παρκώς διαφανείς. Φαίνεται ότι ως συνήθως το Συμβούλιο εξασθενεί τις ε, προτάσεις της ε, Κομισιόν, ειδικά αυτές που το ανησυχούν βεβαίως. Το Συμβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτές τις ε, συστάσεις, αλλά αυτό ευθυγραμμίζεται και με τον νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ε, θεματοφύλακα της ε, λογοδοσίας και της διαφάνειας του Κοινοβουλίου, δηλαδή να βρει τους λόγους για τους οποίους έγιναν κάποιες αλλαγές. Οι επιτροπές θα διοργανώσουν πιο λεπτομερείς ακροάσεις για το θέμα αυτό τον Νοέμβριο, στις οποίες έχουμε προσκαλέσει Συμβούλιο και Κομισιόν. Άλλα ερωτήματα τα οποία θέτει το Κοινοβούλιο αφορούν την διάδραση μεταξύ των αναγκών ε, που έχουν νομική φύση, τα εθνικά προγράμματα τα οποία ακόμα δεν είναι δεσμευτικά, οι συστάσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές, καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης των ε, δεσμεύσεων των κρατών μελών όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όλα αυτά έχουν κρίσιμη σημασία για να ενισχυθεί σημαντικά η οικονομική διακυβέρνηση που χρειάζεται η Ευρώπη ως αποτέλεσμα Τη συνεχόμενη κρίσης. Σας ευχαριστώ κυρία Μπόλ. Σε επόμενη ομιλήτρια, συντάκτρια και αυτή της προφορικής ερώτησης για την, τον ίδιο χρόνο, κυρία Μπερέ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Το Κοινοβούλιο, ε, θέτοντα αυτή την προφορική ερώτηση, θέλει να τη συμπεριλάβει σε μια συζήτηση την οποία κρίνει απολύτω απαραίτητη. Έλαβε η Κομισιόν την πρωτοβουλία να δρομολογήσει την πρόταση αυτή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με την ιδέα στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης ε, ότι πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό ε, για να έχουμε αυτή την περιβόητη τελικά οικονομική κυβέρνηση. Διερωτώμεθα, ε, μπορεί να υπάρχει οικονομική κυβέρνηση χωρίς οικονομικό κοινοβούλιο. Εξού και σας ε, ερωτούμε πώς αξιολογείτε τη δημοκρατική νομιμότητα αυτού του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Πώς θα γίνει ο δημοκρατικός διάλογος γύρω από αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο, πώς θα συζητηθούν οι προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής, γιατί αυτό είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Αν λοιπόν αυξάνεται το επίπεδο στο οποίο γίνεται η διαιτησία των ε, οικονομικών πολιτικών και αποφάσεων, δεν μπορείτε να αγνοείτε την πολιτική συζήτηση και τις πολιτικές αποφάσεις ε, γύρω από αυτούς τους προσανατολισμούς. Εξού και προσπαθούμε ε, ως Κοινοβούλιο να συμμετάσχουμε και γι' αυτό και οι, προσωπικές, οι προφορικές μας ερωτήσεις. Αναφέρατε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καταφέρατε να το κάνετε αυτό χωρίς να αναφέρετε ούτε μία φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και τα εθνικά κοινοβούλια προσθέτω εν παρόδο. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει δεσμευθεί ήδη από το Δεκέμβριο να έχουμε την τελευταία έκθεση για τον ανταγωνισμό. Σύμφωνοι, γιατί δεν συζήτησατε μαζί μα όμω αυτό το θέμα. Πού βρίσκεται η δημοκρατική συζήτηση, ο δημοκρατικό διάλογο, όταν λοιπόν θα υποβάλλετε ε, τη νέα πρόταση, με βάση ποια αξιολόγηση του κύκλου που μόλι ολοκληρώθηκε θα προβείτε σε αυτή την άσκηση. Πώς θα συμπεριλάβετε την εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης 2020 ε, στην ανάλυση αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, όπως είπε και η κυρία Μπόλς και την υποστηρίζω πλήρως και σε αυτό το σημείο και σε πολλά άλλα, ζητούμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τις τροποποιήσεις τις οποίες εσείς επιφέρετε μετά από συζήτηση με τα κράτη-μέλη για τις ειδικέ αναχώρασεις τάσεις. Διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει καμία νομιμότητα αυτό το εγχείρημα και δεν έχει κανένα νόημα. Όταν εγκρίνεται λοιπόν τελικά την αιτήσια έκθεση και εξέταση του ανταγωνισμού, τι σημασία αποδίδεται στο έγγραφο αυτό. Είναι απλά ένα γραφειοκρατικό έγγραφο για να διασκεδάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι ένα πραγματικό έγγραφο προς ανατολισμού. Ελπίζω να μην αυτά και θέλουμε να μας πείτε και τι πιστεύετε για το σύμφωνο Europlus. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπέρες, λέει πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο εκ μέρους ε, του Συμβουλίου στον κύριο Ντομινίκ. Dzień dobry, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας ε, κυρίες ε, και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης ε, να σας ευχαριστήσω τις κυρίες Μπόουλς και Εμπερές, για τις ερωτήσεις που έκαναν. Νομίζω πως είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για να μοιραστούμε μαζί σας την πρώτη μας αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού εξαμήνου και για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τη μελλοντική εφαρμογή του. Θα ήθελα να τονίσω πως ε, πρόκειται για μια αρχική αξιολόγηση γιατί ε, βεβαίως όλες οι σχετικές διαδικασίες του εξαμήνου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον αυτό το πρώτο εξάμεινο όταν τα εθνικά κοινοβούλια υιοθετήσουν ε, τους ε, προϋπολογισμούς τους. Οπότε αυτή είναι όταν ε, θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Τώρα θα δούμε αν έχει υπάρξει κάποια επιπρόσθετη προστιθέμενη αξία στην διαδικασία των Εθνικών Κοινοβουλίων περί του προπολογισμού. Εδώ πέρα αναφέρομαι βεβαίω στην συνέργεια μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών και μια μεγαλύτερη σύγκληση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Η διαδικασία συνεχίζεται και θα πρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όμως, η πρώτη εμπειρία μας λέει πως ε, είναι κάτι το επιθυμητό και μια σωστή διαδικασία την οποία παίρνουν πολλοί στα σοβαρά τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι βουλευτές πώς έχει η διαδικασία. Ξεκινάει τον Ιανουάριο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την ετήσια ανάλυση της για την ανάπτυξη και μετά το ΕΚΟΦΗΝ του Φεβρουαρίου υιοθετεί γενικές κατευθυντήριες γραμμέ για τα κράτη-μέλη και μετά τα κράτη-μέλη έχουν καιρό μέχρι τον Απρίλιο για να συντάξουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα και να προσαρμόσουν τα προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης και μετά βεβαίως υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Μετά έχουμε τις απόψεις των ε, κρατών μελών. όσον αφορά τις ε, τοποθετήσεις αυτές. Και βεβαίως σημαντικότερη περίοδος είναι ο Ιούνιος, καθώς ε, όλα τα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο τελικά υιοθετούν αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, οι οποίες όπως ε, και φέτος επιβεβαιώνονται από το ΕΚΟΦΗΝ. Φέτος ήταν το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών στις 12 Ιουλίου. Είναι λοιπόν πολύ συχτό και πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε κάποιες προτάσεις για να βελτιωθεί η διαδικασία. Θα ήθελα όμως να σας πω πως η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να γίνεται με δύο ε, πτυχές. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ε, επιχειρησιακή πτυχή, τις διαδικασίες δηλαδή με τις οποίες ε, υιοθετούνται οι αποφάσεις και το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στον πολιτικό διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάμειξη των κρατών μελών και βεβαίως τον αντίκτυπο που έχει στα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλουμε λοιπόν να συνδυάζουμε μακροοικονομικές ε, προτεραιότητες με τις δυνατότητες που υπάρχουν στα δημόσια οικονομικά όσον αφορά την πρώτη πτυχή, την καθαρά τεχνική. Μετά από τους μήνες αυτούς ε, και την διαδικασία την οποία ανέλησα για τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, μπορούμε να πούμε πως ε, είναι εξαιρετικά τεχνική η διαδικασία και απαιτεί πάρα πολλά έγγραφα καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της αλληλογραφίας που συνεχίζεται επί έξι μήνες. Μιλάμε για 600 περίπου έγγραφα τα οποία πρέπει και να μεταφραστούν σε επίσημες γλώσσες οπότε και από τεχνική σκοπιά είναι περιπλοκή διαδικασία. Κατόπιν το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό, δηλαδή ειδικά τον Ιούνιο οι προθεσμίες είναι πάρα πολύ πιεστικές για να υιοθετηθούν αυτά τα έγγραφα αφού υιοθετηθούν πρώτα απ' όλα οι συστάσεις και μετά δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στη φάση αυτή. Οπότε προκύπτει το ερώτημα του πώς θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Μία από τις προτάσεις η οποία προκύπτει από την εμπειρία που είχαμε και ελπίζω έτσι να γίνουν τα πράγματα στο μέλλον είναι πως θα ξεκινήσει μάλλον νωρίτερα η διαδικασία και θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την αρχική της έκθεση ήδη τον Δεκέμβριο. Έτσι θα έχουμε κάποιες εβδομάδες παραπάνω για να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, οπότε να μπορούμε τον Απρίλιο να έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο όταν ε, πρόκειται για τις απαντήσεις ε, των κρατών μελών στις προτεραιότητες που αναφέρει η έκθεση της ε, Κομισιόν. Και μετά βεβαίως θα συντάσσονται τα έγγραφα τα οποία αφορούν το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη ή τα εθνικά, μεταρθυστικά προγράμματα. Έτσι θα μειωθεί η πίεση και η ένταση η οποία κορυφώνεται τέλος Μαΐου και τον Ιούνιο για να συντονιστούν αποτελεσματικά όλα αυτά τα θεσμικά όργανα και να υιοθετηθούν όλες αυτές οι προτάσεις. Θα ήθελα επίσης να ευστήσω την προσοχή σας στην αποφασιστικότητα των κρατών μελών για να είναι αποτελεσματικά ήδη φέτος. Όπως σας είπα, πρόκειται περί 600 εγγράφων, πολύ πιεστικές προθεσμίες, οπότε τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να αποκλίνουν ε, από τις ε, συνήθεις ε, διαδικασίες και να συζητήσουν έγγραφα παρά το ότι δεν ήταν μεταφρασμένα κάτι το οποίο συμβαίνει σπάνια αλλά δείχνει το πόσο μας απασχολούσε αυτή η διαδικασία. Εργάστηκαν με αγγλικά ή γαλλικά κείμενα για να επιταχυνθεί η διαδικασία για να μπορέσουν να υιοθετηθούν όλες οι συστάσεις εγκαίρως. Τώρα θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικότερο πρόκειται για την αξιολόγηση του αντικτύπου στο, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον οικονομικό διάλογο. Πρέπει να θυμόμαστε πως ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μόνο ένα στοιχείο μεταξύ ενός φάσματος ε, εργαλείων ε, τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέα μέσα για να ενισχυθεί η οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να έχουμε καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Έχουμε το εξαπλό πακέτο, όπως ξέρετε, έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, έχουμε και την συνήθη, θα έλεγα, εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν ε, περισσότερη διαφάνεια και ενισχύουν ε, τον διάλογο μεταξύ των ε, κρατών μελών. Η διαφάνεια επίσης ενισχύεται όσον αφορά την πραγματική οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη καθώς ε, αυξάνεται και η πίεση στα κράτη-μέλη για να γίνει η συζήτηση με σωστό τρόπο και για να μπορέσουν όλοι να έχουν ε, μία ιδέα του πού οδεύουμε ως ε, Ένωση. Οπότε, από πρακτική σκοπιά, αυτό το οποίο εισήχθη με το εξαπλό πακέτο ήταν το εξής. Πρώτα απ' όλα, μια μεγαλύτερη και καλύτερη ανάμιξη των εθνικών κοινοβουλίων στην διαδικασία της ε, μεταφοράς ε, των προτεραιοτήτων της Ένωσης και της μετατροπής τους σε εθνικές ε, προτεραιότητες μέσω του ισχυρότερου δυνατού μέσου, δηλαδή του εθνικού προϋπολογισμού. Οπότε αυτή τη στιγμή τα Εθνικά Κοινοβούλια ενημερώνονται για τις ε, προτεραιότητες οι οποίες ε, θα προταθούν από, ένα κράτος, από το κάθε κράτος μέλος στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και το τι σημαίνει αυτό για τον ε, προϋπολογισμό τους. γιατί αυτό αποστέλλεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά βεβαίως ε, υπάρχουν ε, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και μετά τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν τον τελικό λόγο όσον αφορά τη διαμόρφωση του εθνικού προϋπολογισμού. Δηλαδή υπάρχει ένα μέσο ελέγχου του πώς ε, οι προτεραιότητες και οι στάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταφράζονται στην ε, πράξη. Οπότε υπάρχει μια ενίσχυση της κοινή κατεύθυνση όλων των κρατών μελών, εάν η προτεραιότητα είναι να διατηρηθεί, να ενταθεί η ανάπτυξη σε κάποια κράτη-μέλη η εφαρμογή του προγράμματος για το 2020. Αυτό τονίζεται σαφώς, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Οπότε δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο το οποίο θα εφαρμόζουν όλοι. Έχουμε μεμονωμένες συζητήσεις των κρατών μελών που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του καθενός και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως τα μέσα τα οποία θα υιοθετηθούν είναι θέμα των κρατών μελών ταυτόχρονα. Υπάρχει καλύτερος ε, συντονισμός και πιο στοχευμένη χρήση των ευρωπαϊκών πόνων γιατί τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας και ορίζουν το ποιους ε, στόχους ε, στηρίζουν ε, με τα κονδύλια τα οποία λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως αυτό συνδέεται με άλλα προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων. Οπότε έχουμε κατόπιν τις ε, Έχουμε τις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τις χρηματοδοτήσει και θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να προσανατολίσουν τις δαπάνες του προπολογισμού προς αυτή την κατεύθυνση. Το μήνυμα είναι σαφές. Οπότε νομίζω πως ε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το ευρωπαϊκό εξάμεινο ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι το πώς θα μεταφραστεί στους εθνικούς προπολογισμούς γιατί αυτό όπως είπα επαφίεται στα εθνικά κοινοβούλια αλλά έχουμε τα μέσα, τις δυνατότητες στη διάθεσή μας και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και βεβαίως μπορεί η τελική μας αξιολόγηση μετά το τέλος του έτους να περιέχει συστάσεις για το τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Και βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει μια μεγάλη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τον τραπεζικό τομέα. Οπότε η οικονομική κατάσταση της Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται δυναμικά αυτό το οποίο θεωρούσαμε εμείς ε, προτεραιότητες τον Απρίλιο ή τον Μάιο οι στόχοι τους οποίους θα μπορούσαμε να επιτύχουμε με βάση τα δεδομένα της άνοιξης της ε, φετινής ε, μπορεί να αποδειχθεί αδύνατο να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή ή να μην επαρκεί. Οπότε μάλλον σε λίγες εβδομάδες θα ακούσουμε κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες θα λένε πως παρά το ευρωπαϊκό εξάμεινο οι στόχοι δεν έχουν ε, επιτευχθεί, αλλά βεβαίως η εξέλιξη της κρίσης ε, είναι δυναμική, οπότε είναι δύσκολο να προβλέψουμε όλες ε, τις δράσεις που θα έπρεπε να αναλάβουμε. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το εξαπλό αυτό πακέτο είναι μέσα τα οποία έχουν στόχο να μας βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι τα μέσα τα οποία θα ξεπεράσουν ε, την κρίση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πως μόνο με την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού εξαμήνου θα έχουμε αυτομάτως καλύτερη οικονομική κατάσταση στην Ένωση, αλλά κατά την άποψή μας η ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Εξωμήνου βελτίωσε το μακροοικονομικό διάλογο στην Ένωση και αυτός ήταν ο βασικός στόχος. Οπότε η πρώτη αξιολόγηση του Συμβουλίου όσον αφορά την, την ε, διαδικασία ήταν αυτή και προσπαθούμε βεβαίως να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς θα βελτιωθεί και πώς θα εμπλακούν ακόμη καλύτερα τα κράτη-μέλη και πώς θα βελτιωθεί ο διάλογος, όπως σας είπα, για τις ε, συστάσεις. Και όσον αφορά την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, διαδικασία, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι διαφανής, όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες, δημοσιεύονται, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση και έλαβε μέρος στην ε, διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκάλεσε εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συζητήσουν. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας ε, την εκτίμησή μας για αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο καθώς και τα σχέδιά μας για τον επόμενο χρόνο. Το πρώτο ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της οικονομικής μας διακυβέρνησης. Ε, αποτελεί τμήμα μιας προσπάθειας για την ανανέωση της εμπιστοσύνης με σωστή εστιασμό στην κατασκευή των θεμελίων για την απασχόληση και την ανάπτυξη και για να ενισχυθεί ο σχεδιασμός, πολιτικός σχεδιασμός και η εφαρμογή αυτού. Είχαμε σαφείς προσδοκίες για το τι θα έπρεπε βασικά να επιτύχει επί της ουσίας το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Καταρχήν θέλαμε να εξασφαλίσουμε στενότερη συνεργασία για την ανάλυση, την πολιτική και τις οδηγίες για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές αλλά και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Δεύτερον, θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές κατευθύνσεις που δίνονται στα κράτη-μέλη θα είχαν μεγαλύτερη επιρροή για την εφαρμογή, για καλύτερο συγχρονισμό των πολιτικών αυτών κατευθύνσεων και ε, θα οδηγούσαν σε πιο συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έπρεπε να εξασφαλίσει ότι η διάσταση της Ένωσης όσον αφορά την, ε, την πολιτική και τον αντίκτυπο αυτής θα, θα λαμβανόταν εξ αρχής υπόψη. θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ήταν επιτυχές το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε αυτά τα σημαντικά ε, στοιχεία. Όσον αφορά την αξιολόγηση των ε, εκ των προτέρων πολιτικών κατευθύνσεων και την ε, συνέχεια που δίνουν τα κρατημένα, είναι κάπω νωρί για να πούμε τι έγινε, γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε στα μέσα του εθνικού εξαμήνου και θα μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση όταν οι προπολογισμοί των κρατών μελών καθώς και οι διευθυντικές αλλαγές θα έχουν αποφασιστεί και θα τις έχουμε και αξιολογήσει και βεβαίως ε, υπολογίζω στο σώμα σας ότι θα μας βοηθήσετε στην αξιολόγηση. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια ποιο θα είναι ο αντίκτυπο των μέτρων που θα έχουν ληφθεί. Υπάρχει, αναγνωρίζεται από όλου του εμπλεκόμενου φορεί ότι οι πολιτικέ κατευθύνσει είναι πιο ολοκληρωμένε σε διάφορου ε, πολιτικού τομεί με εστιασμό περισσότερο στις χώρες και στις προτεραιότητές τους. Επίσης είναι πιο εύκολη η εφαρμογή τους. Με την κοινή παρουσίαση των ε, κατευθυντηρίων αυτών ε, πολιτικών καθώς και των εθνικών πολιτικών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα βασικά πολιτικά προγράμματα ε, τα οποία έχουμε, τα έχουμε εξετάσει και έχουμε προτείνει πολιτικές συστάσεις με βάση το, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως νομικό μέσο. Έχουμε δε εξασφαλίσει πως τα εθνικά προγράμματα θα λαμβάνουν υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση εξ αρχής. Ενώ θεωρώ λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι σαφώς επιτυχές και σημαντικό βήμα προόδου, υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτίωση. Το 2012 το πιο πιο σημαντική πτυχή θα είναι ισχυρότερος εστιασμός στην διάσταση της ανάπτυξης. Όπως ε, το τόνισε στις 12 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Μπαρόζο, η ανάπτυξη εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή των βασικών μεταρρυθμίσεων στην εσωτερική αγορά, αλλά και από τα νέα δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα, τα ομόλογα έργου που θα βοηθήσουν να εξέλθει η Ευρώπη από την κρίση. Η Κομισιόν επίσης αποφάσισε να, να κάνει την ε, παρουσίαση της έρευνας για την εφαρμογή του εξαμήνου στα τέλη του 2011, νωρίτερα δηλαδή από ό,τι προβλεπόταν, γιατί όλα αυτά μπορούν να στηριχθούν ε, μέσω νομιμότητας όταν αυτά είναι σωστά αγκιστρωμένα στη δημοκρατική διαδικασία, καθώς ε, και εφόσον θα αποδώσουν ε, και θα εξυπηρετήσουν ε, το κοινό καλό. Αυτό σημαίνει βέβαια πως το, το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ισχυρός δεσμός ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Διάσταση και την Εθνική Διάσταση για τις βασικές ε, πολιτικές προκλήσεις μπορεί να θεσπιστεί μόνο αν αυτές οι προοπτικές ε, συνδυαστούν και αυτό θα γίνει μόνο αν τα κοινοβούλια παίξουν ισχυρό ρόλο. Πιστεύω ότι στην αερινή διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που εσεί διοργανώσατε το 2011 θα μπορούσε να επαναληφθεί και να αποτελέσει ένα σημαντικό θεσμικό τρόπο για καλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και εξασφάλιση τη νομιμότητα. Βεβαίω, η νέα νομοθεσία περί οικονομική διακυβέρνηση υπογραμμίζει την ανάγκη τα Εθνικά Κοινοβούλια και άλλοι φορεί να συμμετέχουν πλήρω στο εξάμεινο, καθώ και στην επεξεργασία των ε, ε, SCP και των NRP. Εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Γκοζέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Σημειώνω στα λόγια του Επιτρόπου ότι ήταν επιτυχέ ε, το εξάμεινο και αυτό με ικανοποιεί τη στιγμή που βιώνει η Ευρώπη μια δραματική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο, όπως το αποκαλούμε, να ε, επιτύχει κάποια ε, πρόοδο. Θα ήθελα να στραφώ όμω στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Για 16 λεπτά ε, προσπαθούσατε να μα εξηγήσετε ε, ένα μηχανισμό τον οποίο γνωρίζουμε και μα είπατε ότι είναι πολύ τεχνικό. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και ότι αν θέλουμε να ενημερωθούμε έχουμε τύχη γιατί μπορούμε στο διαδίκτυο να βρούμε τα έγγραφα τα οποία δημοσιοποιούνται για όλους. Μήπως ε, θα μας πείτε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες, κάτι που κάνουμε καθημερινά. Εμείς σας ρωτήσαμε ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εσείς μας απαντήσατε, διαβάστε τις εφημερίδες και δείτε στο διαδίκτυο Εμάς ξέρετε μας ρωτάνε τι κάνει η Ευρώπη σε, αυτές τις, ε, ε, σε αυτή την κρίση ε, και λέμε ότι ορίστε έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τελικά όμως το ευρωπαϊκό εξάμεινο τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια μέθοδος που θα βοηθήσει την Ευρώπη να εξέλθει από την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζές. Κύριε Ποδηματά, τώρα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εξ αρχής είχε υποστηρίξει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θεωρώντας ότι υποτελεί μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία που έχει στόχο την έγκαιρη ευθυγράμμιση των εθνικών προπολογισμών και των προγραμμάτων διαρθρωτικών αλλαγών, όχι με τους στόχους της Ένωσης γενικώ, αλλά ειδικότερα με τους στόχους ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας για να κάνουμε όμως ε, έγκαιρα τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις χρειάζεται να ε, αντλήσουμε ορισμένα συμπεράσματα από την πρώτη εφαρμογή αυτής της διαδικασίας και κατά την πρώτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού εξαμήνου είχαμε ένα μάλλον περιορισμένης κατεύθυνσης κείμενο ουσιαστικής απόκλισης των κρατών μελών από τους στόχους ανάπτυξης βάσει της στρατηγικής ευρώπη 2020 αλλά και μη τήρησης ορισμένων συστάσεων της επιτροπής ανά κράτος μέλος με πρωτοβουλία του συμβουλίου. επειδή εκείνο που φαίνεται να εξελίσσεται το είπαν και άλλοι συνάδελφοι σε βασικό πρόβλημα της ένωσης στην παρούσα κρίση είναι οι καθυστερήσεις η μη έγκαιρη εφαρμογή των αποφάσεων και κυρίως η έλλειψη συνοχη μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ένωσης θέλουμε να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο να επιμείνουμε δηλαδή ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου χρειάζεται μια ουσιαστική και περιεκτική πρόταση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη και η πλήρης εφαρμογή της κοινοτικής διαδικασίας με εμπλοκή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αποδηματά. Η Σιλβί Γκουλάρ τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Γκοζές ε, θέλω να σας πω σε ποιο πλανήτη ζείτε κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Σε ποιο πλανήτη ζείτε. Ο Επίτροπο βέβαια μίλησε με μεγαλύτερη επίγνωση για την ανάγκη δημοκρατική νομιμότητα των αποφάσεων σε οικονομικά θέματα, αλλά σα ρωτώ και εσά κύριε Επίτροπε, συζητάτε με άτομα που βρίσκονται στο μάτι του κυκλών αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ε, πώ μα αντιλαμβάνεται ο κόσμο. Μήπω ε, δεν θα έβλαπτε και λίγη αυτοκριτική. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία, ξεκίνησε, αλλά είναι ανεπαρκέστατη. Εγώ θα επιμείνω σε ένα σημείο. Με κάθε ειλικρίνεια προσβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το να μας λέτε πηγαίνετε και δείτε στο διαδίκτυο και έτσι θα έχετε συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό προσβάλλει τη δημοκρατία. Δεν θέλουμε ζητιανιές και επαιτία για ενημέρωση. Θέλουμε πληροφορίες συγκεκριμένε, οικονομικές, ε, κοινωνικές, φορολογικές, πολιτικές. Πολύ σημαντικές αλλαγές θα γίνουν. Θέλουμε να έχουμε ενημέρωση για αυτές τις πολιτικές που θα βοηθήσουν ε, να ε, βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειαζόμαστε κινητοποίηση των Εθνικών Κοινοβουλίων, χρειαζόμαστε γενική κινητοποίηση και λίγο περισσότερη ενημέρωση και διαβούλευση και κάτι παραπάνω. Μια διασυνοριακή συζήτηση και το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ένα από του χώρου που θα γίνει αυτό ο διάλογο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στρέτσεκ, για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή την ομιλία του εκπροσώπου του Συμβουλίου και σίγουρα θα είμαι ο μόνος εδώ που θα πω ότι είμαι ικανοποιημένο από αυτή την ομιλία γιατί το Συμβούλιο τοποθετείται μέσα στον πραγματικό οικονομικό χώρο. Μάλιστα αυτό μας είπε και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια και η συζήτηση στο πλαίσιο των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν είναι καθόλου εύκολη και δεν είναι και μονόδρομοι. Ε, μας περιγράψατε μια ξεκάθαρη αλήθεια ότι δηλαδή οι εθνικές οικονομίες αμφισβητώνται και η εναρμόνισή τους δεν μπορεί να γίνει εν μία ανοιχτή. Εφόσον το Συμβούλιο λοιπόν μας λέει ότι πρόκειται για 600 έγγραφα τα οποία μάλιστα δεν είναι όλα σε εθνική γλώσσα τότε τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει και αυτά να κινητοποιηθούν και αυτό απαιτεί χρόνο. Και βέβαια όλα αυτά δεν αντιστοιχούν στις οικονομικές αναταράξεις της, ε, της πραγματικής οικονομίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας ε, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον κύριο Επίτροπο φαίνεται πως είναι μεγάλη επιτυχία το εξάμεινο αυτό. Έχω τις αμφιβολίες μου. Εάν δούμε τις συστάσεις που έγιναν στα κράτη-μέλη όλες αυτές ακολουθούν μία γραμμή. Κοιτάμε μόνο τις δημόσιες δαπάνες και εκεί πέρα πρέπει να γίνουν όσο δυνατόν περισσότερες οικονομίες. Αυτή είναι η βασική γραμμή αν δει κανείς συστάσεις της ο κύριος ε, Νταλή μας λέει πως την επόμενη φορά θα δούμε και την απασχόληση. Είναι μια βελτίωση αυτή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του εξαμήνου. Θα πρέπει να συνεισφέρει το εξάμεινο στρατηγική 2020 και έχετε πέντε κυρίους δείκτες. Έρευνα, απασχόληση, εκπαίδευση, καταπολέμηση της στόχιας και περιβάλλον. Αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είναι τα βασικά και θα έπρεπε να φαίνονται στις συστάσεις. Είδαμε λοιπόν όλους ε, τους διαφόρους δείκτες και βλέπουμε πως η Κομισιόν έχει κάνει συστάσεις που δεν κολλάνε με αυτούς τους στόχους. Ένα παράδειγμα, ε, εξοικονόμηση της, ερεύνη, της ε, ενέργειας, πάρα πολύ σημαντικό ε, έχουν κάνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν τα αναφέρει καν η Κομισιόν. Άλλο ζήτημα, έρευνα. Από 3% πήγε 2,5%. Και τι μας λέει η Κομισιόν, ε, και το 2,5% καλό είναι. Δηλαδή δεν έχει σημασία ο στόχο του 3%, τότε πείτε το. Εάν είναι αυτή η γραμμή της Κομισιόν, τότε πείτε το και ξεκάθαρα πως η ατζέντα του 2020 δεν έχει πια καμιά σημασία και κοιτάμε μόνο τους οικονομικούς δείκτες. Να είστε τουλάχιστον ειλικρινείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι στόχοι αυτοί αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα πρέπει να κοιτάτε όλους τους δείκτες ή αλλιώς να είστε ειλικρινείς και να ξεχάσετε αυτή την ατζέντα για το 2020. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει ο κύριος Χουντής για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι απαντήσεις των εκπροσώπων του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν ε, στην ερώτηση των συναδέλφων ουσιαστικά εμφάνισαν το πρόβλημα ως ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Όμως αγαπητοί συνάδελφοι το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι εξόχως πολιτικό. Κατά την άποψή μου η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι αντικοινωνική, αντιδημοκρατική, αντιδραστική καθώς τα κράτη μέλη κάτω από τις πολιτικές πιέσεις και τις απειλές της κομισιόν προσαρμόζουν τους δημοσιονομικούς τους στόχους προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς. με την εφαρμογή ουσιαστικά αφαιρείται κάθε δυνατότητα από κάθε κράτος μέλος ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση έχει ψηφίσει να εφαρμόσει αφαιρείται αυτή η δυνατότητα εναλλακτική αναπτυξιακή πολιτική. αντιθέτως ανεξάρτητα από ποια πολιτική ενέκρινε ο λαός κάθε χώρας πρέπει να εφαρμόζει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας της ευρωπαϊκής ένωσης τελικά αν στην ελλάδα ο άνεργος πάρει επίδομα ανεργίας αν στην ιρλανδία ο φτωχός και ο άστεγος θα έχει παροχές πρόνοιας αν στην πορτογαλία ο εργαζόμενος παίρνει 300 ευρώ θα το αποφασίσει ο κύριος Μπαρόζο ή ο εκάστοτε κύριος Μπαρόζο ή ο εκάστοτε κύριος Ρεν. Τέλος, αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μια νομιμοποίηση όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση που παραβιάζει τις συνθήκες της ευρωπαϊκής ένωσης που παραβιάζει και παρακάμπτει τα εθνικά κοινοβούλια που παρακάμπτει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και κυρίως που παρακάμπτει και παραβιάζει και παραβλέπει τα συμφέροντα των λαών. κύριε επίτροπε κύριε του συμβουλίου αγαπητοί συνάδελφοι τούτε τις ώρε που λαμβάνονται ή θα ληφθούν από του ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον έλληνα πρωθυπουργό αποφάσει για τη διαχείριση του χρέους αυτές οι αποφάσεις αν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση τότε δεν φτάνουν τα ευρωπαϊκά εξάμενα για να σώσουν την κατάσταση. αντιστρόφως θα ζήσουμε ένα εκρηκτικό πανευρωπαϊκό εξάμεινο από τις κινητοποιήσεις των ευρωπαίων εργαζομένων που θα πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ο κύριος ε, απουσιάζει από βλέπω. Άρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βέχτμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα μέσο πολιτικής κατεύθυνσης για να ενισχυθεί η στρατηγική του 2020. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη την Άνοιξη να παρουσιάσουν τα οικονομικά του σχέδια, κάτι το οποίο κρίθηκε αναγκαίο για να αντιμετωπιστεί η καταστροφική οικονομική κατάσταση πολλών κρατών μελών. Εδώ πέρα θα ήθελα να πω πως συμφωνώ με την τεχνική κριτική των συναδέλφων. Η εξάντληση της δυναμικότητας της ε, κοινή αγοράς ε, είναι ένας από τους δέκα στόχους ε, της ε, έκθεσης 2011 που θα πρέπει να γίνει μέχρι το 2012. Απαιτείται από όλους μας να ενισχύσουμε αυτό το δυναμικό μέσω χρηματοδότησης ε, έργων υποδομής και αύξησης της ε, ανταγωνιστικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας για να δημιουργηθεί ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία ο κύριος Μπάλτς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, από ό,τι φαίνεται συμφωνούν μαζί μας καθώς υπογράμμισαν την ε, Κυριακή πως ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Μίλησαν μάλιστα και για μαθήματα του παρελθόντος. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχει ήδη μια εμπειρία την οποία είχαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Συμφώνου Σταθερότητος. Ο αυτοέλεγχος του Συμβουλίου δεν λειτουργεί, δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Οπότε είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε κάποιες μεγάλες δημόσιες παραδοχές στον τομέα της, ε, του συντονισμού και να τα εφαρμόσουμε κιόλας. Τελικά καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Θα πρέπει να ενισχυθεί το σύμφωνο σταθερότητα, αλλά αυτό δεν επαρκεί. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινοτική μέθοδο, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μια ανοιχτή συζήτηση για τι ετήσιε εκθέσει ανάπτυξη, για τι συστάσει κομισιών και για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αλλά η μεγάλη ευθύνη εξακολουθεί να υπάρχει στην Κομισιόν. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες βελτίωσης που υπάρχουν γιατί βεβαίως δεν αρκεί να δημιουργήσουμε ένα νέο μέσο, πρέπει να το χρησιμοποιούμε και αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Για ένα λεπτό αν και είναι νωρί όπως υπόθηκε για οριστική απόφαση, είναι δύσκολο κανείς να μην έχει την άποψη ότι αυτό το εξάμεινο προκαλεί έναν αδύναμο συντονισμό και μια αμφίβολη δημοκρατική νομιμότητα και αυτά τα θέματα συνδέονται γιατί χωρίς δημοκρατική νομιμότητα περισσότερο πρόκειται για γραφειοκρατική υπόθεση και όχι για ουσιαστικό συντονισμό. Ε, μιλήσατε για τις αρχές του Κοινοβουλίου, για τις, ε, για τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου που θα έπρεπε να αποτελεί τον κόμβο για αυτήν την ε, ε, προσπάθεια. Θα έπρεπε ωστόσο άμεσα να χρησιμοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί που προβλέπονται από τη συνθήκη για να ενισχυθεί η συνεργασία και να δοθεί μεγαλύτερο ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, ε, Διαβάζοντα τι συστάσει του Συμβουλίου, φαίνεται να υπάρχει ένα προφανέ όριο τη οικονομική γραμμή που τη έχει πνευεί. Μείωση, μείωση του ελλείμματο, ναι, απαραίτητε προποθέσει, αλλά όχι επαρκή για να αντιπαρέλθουμε την ε, κρίση. Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε έναν φαύλο κύκλο που θα μας ε, ε, κατευθύνει προς την κατάρρευση. Είναι αντικείμενο μιας γνήσιας πολιτικής συζήτησης που δεν μπορεί παρά να γίνει παραμέσω διαλόγου ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Γκουαλτιέρη, ο κύριος Χάγκλοντ για μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως ε, όταν μιλάμε με τον κόσμο μας ρωτάνε γιατί ασχολείστε με τα δομικά και τα διαστατικά στην Ευρώπη και δεν λύνετε την κρίση. Συζητάμε για θεσμικά και όχι για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Λέγεται πως η κρίση ε, μπορεί να λυθεί με τα εργαλεία τα οποία έχουμε. Πριν από ένα μήνα εγκρίναμε το λεγόμενο εξαπλό πακέτο και ακούσαμε πως ε, μέρος αυτού βεβαίως αποτελεί και το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα αυτό σκεφτόμαστε αντί να το εφαρμόσουμε στα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε. Ναι, πράγματι χρειαζόμαστε μια γενική δημόσια συζήτηση και γι' αυτό είναι εδώ πέρα το, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν κάνει και τις ε, συστάσεις της, αλλά δεν νομίζω πως ε, ε, μας βοηθάει και σε τίποτα αυτή τη συζήτηση. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Ε, ακούστηκαν πολλά έξυπνα πράγματα για το τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την ανάπτυξη. Η οικονομία, μόνο η εξοικονόμηση δεν θα μας βγάλει από την κρίση. Ναι, πρέπει βεβαίω να εξοικονομήσουμε, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να σκεφτούμε πως ε, πρέπει να έχουμε μια νέα σειρά εργαλείων για τη λύση της κρίσης. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες στους οποίους εκπροσωπώ ίσως και να μην ενδιαφέρονται κατά ανάγκη για το τι συμβαίνει σε ένα απομακρυσμένο ευρωπαϊκό εξάμενο, αλλά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της, ότι επιδεινώνεται η κρίση. Πολλοί πολίτες μας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πουχτήσει που πρέπει να διασώσουν συνέχεια τις ε, τράπεζές τους. Ε και ταυτόχρονα βλέπουν ε, τις ε, τράπεζες στην ε, υπηρετική Ευρώπη να πρέπει να αναδιαρθρωθούν. Είναι πολύ επώδυνες όλες αυτές οι καταστάσεις. Εγώ τώρα σε ό,τι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θεωρώ και ελπίζω να αρθούν στο ύψος των προσδοκιών τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ε, την συγκεκριμένη οδηγία πλαίσιο, γιατί θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει πού πηγαίνουν τα χρήματα των φορολογμένων, πώς δαπανώνται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μία από τις πρώτες δράσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του επόμενου έτους θα πρέπει να είναι ε, τα κράτη-μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Ευχαριστώ κύριο Σμέλτζερ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, με το να μεταφερθούν τα θέματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον δεν μπορούν οι αγορές να επιβάλλουν την πειθαρχία τους. Αντί παραδείγματος χάρη να δώσουμε την ευκαιρία στους Έλληνες ε, να ανακάμψουν, ε, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να διευκολύνουμε την υπερχρέωση Επίσης έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκή εποπτεία των προϋπολογισμών αλλά θα καταλήξουμε σε μια γραφειοκρατία κεντρικού σχεδιασμού και το να οδηγήσουμε βεβαίως ε, σε μια τέτοια κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία έχουμε δει σε τι έχει οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε τα βουνά από βούτυρο και τις λίμνες από γάλα. Από ό,τι φαίνεται οι Βρυξέλλες δεν θέλουν να δουν πως η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν μια λανθασμένη κατασκευή η οποία ευθύ εξ αρχή, ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Αντί για περισσότερο συγκεντρωτισμό πρέπει να πάμε ξανά στα ίσα δικαιώματα των κρατών και στην δυνατότητα του καθενός να ορίσει την οικονομική του πολιτική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Τίσεν για λεπτό κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα σχέδια εξαρτώνται από το πώς θα εκτελεστούν. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει κάποια ικανοποίηση για το ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το λεγόμενο six-pack. Αλλά μπορούν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα βήματα όσον αφορά την απαραίτητη οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν υπάρχει εδώ πέρα το απαραίτητο βάρος. Επίσης δεν παρακολουθούνται αρκετά γρήγορα τα γεγονότα και διαπιστώνουμε πως πάρα πολλά κράτη-μέλη πλέον προβάλλουν μεγαλύτερη αντίσταση στον συντονισμό αυτών. Το δεύτερο μέρος ε, της κριτικής αφορά την έλλειψη δημοκρατικής νομοποίησης. Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή μου έχει φτάσει η στιγμή για να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα εφαρμόσουμε την επικουρικότητα ε, ούτως ή άλλως έχουμε καταλήξει σε κάποια ανυπέρβλητα εμπόδια τα οποία πρέπει να αρθούν. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία έχουν ε, υποσχεθεί και θα πρέπει επιτέλους να δεσμευτούν τώρα στο σύνταγμά τους για να διατηρούν ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς. Δεύτερον, πως τα εθνικά κοινοβούλια να δεσμευτούν ρητός για την τήρηση αυτών των ε, δεσμεύσεων και να πάρουν στα σοβαρά την Ευρώπη 2020 και τρίτον συμφωνώ με την περαιτέρω δραστηριοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί χωρίς δημοκρατική νομοποίηση δεν μπορούν να υπάρξουν σοβαρά μέτρα. Ευχαριστώ κυρία Τίσεν. Ο κύριο Κούτα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπα... των... των ευρωπαϊκών κρατών, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή μιας ε, ε, στέρεης οικονομικής διακυβέρνηση. Η οικονομική πολιτική θα έπρεπε να είναι κοινό... ένα κοινό πεδίο δράσης μέσω των ε, προγραμμάτων μας, ε, των εθνικών και των ευρωπαϊκών, θα πρέπει να εγγυηθούμε την ανάπτυξη παιδεία δωρεάν για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και βέβαια δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι συστάσεις προς τα κάτι μέλη θα πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξες ώστε να, μπορεί, να μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020. Αυτή η πρώτη απόπειρα, η πρώτο, ευρωπαϊκό εξάμεινο θα οδηγήσει σε ανάλυση από, τις, από πλευράς της Κομισιόν για την απόδοση των κρατών μελών. Η Κομισιόν θα χρειαστεί να αποφασίσει αποφασίσει μάλλον για τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν από εδώ και μπρος. Ε, βέβαια όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν παρά μόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίξει ρόλο σε όλα αυτά σύμφωνα με την συνθήκη περί λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κούτας. Το λόγο έχει ο κύριος Σμιτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επί της αρχής είμαι θετικός όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ταρχίας και του συντονισμού. Όμως η διάσκεψη κορυφής στην Κυριακή πρότεινε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το Eurogroup. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση 27 κρατών μελών. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν επί ίση όρη. Και αν είναι πάλι να χωριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για μια πορεία επικίνδυνη και λανθασμένη. Και εμείς έχουμε συζήτηση ε, από ό,τι φαίνεται για ένα διαχωρισμό σε χώρε τη Ευρωζώνη και μη βεβαίω αντιλαμβάνομαι το ότι κάτι θέλουν να κάνουν οι χώρες Ευρωζώνης, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην την διαχωρίσουμε και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κυρία Πρόεδρε, η οικονομία μας και στα 27 κράτη-μέλη είναι στενά συνδεδεμένη μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ, κύριος Μπρόνς. Thank you. Η κρίση είναι συμφορά για τους απλούς ανθρώπους, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ευκαιρία για να επεκτείνει τις, αρμο... εξουσίες και τις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμών ε, και να προχωρηθεί προγράμματα όπως η Οικονομική και η Πολιτική Ένωση. Είναι υπερβολική αυτή η συμπεριφορά. Η Οικονομική Πολιτική δεν αφορά τη συμμετρία ή την ομοιομορφία, αλλά τις συγκεκριμένες ανάγκες των διαφόρων οικονομιών. Τα μεγάλα ελλείμματα στους προπολογισμού θα πρέπει πρέπει να αποφεύγονται, αλλά υπάρχουν περιστάσεις υπό τι οποίε είναι ίσω απαραίτητοι. Τώρα, μπορεί να είναι απαραίτητη η η ποσοτική χαλάρωση, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Πάντως θα πρέπει να, δεν μπορεί να επιβάλλεται εξωτερική πειθαρχία που θα επιβάλλει καλές οικονομικές ε, ε, συνήθειες. Σε πόσο καιρό θα πάρει πριν η Κομισιόν αποφασίζει τον προπολογισμό κάθε κράτους μέλους με, και τα κράτη-μέλη να παίζουν απλό συμβουλευτικό ρόλο. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φέιο για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, Καλά έκαναν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν αποφάσισαν ε, την ε, ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι πολύ σημαντικό ο συντονισμό των ε, δημοσιονομικών πολιτικών μαζί με το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Αλλά αυτή η ιδέα αντιμετώπισε πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την εκτέλεσή τη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο απαιτεί πραγματικό συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν το Ευρωκοινοβούλιο Απλά να ενημερώνεται και ίσα ίσα να ενημερώνεται από το ίντερνετ. Οι πολίτες δεν ψήφισαν ευρωβουλευτές που είναι απλά διευθύνσεις ενό email. Ε, ψήφισαν εκπροσώπους των συμφερόντων τους. Και αυτό είναι το πρώτο δίδαγμα που θα πρέπει να αποκομίσουμε. Αλλά κατά δεύτερο λόγο το ευρωπαϊκό εξάμεινο ήδη προχώρησε περισσότερο. Ε, πέτυχε αυτά που είχε πρόθεση να πετύχει. Όχι. Χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σημαντική απάντηση στη σημερινή κρίση. Και εδώ, αν δει κανεί τα νέα ε, τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ ανησυχητικά. Με κάθε ε, ειλικρίνεια, εγώ ε, ε, βλέπω ότι υπάρχει αναποφασιστικότητα και γίνεται λόγο διαρκώ για μελέτε επιμελετών. Δεν χρειαζόμαστε άλλε μελέτε. Χρειάζονται αποφάσει για μια οικονομική κυβέρνηση αποτελεσματική που θα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο, που θα αποφασίζει και θα σκέφτεται για όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Φέιο. Ο κύριο Λούντφιξον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ήδη ακούστηκε στην συζήτηση, δηλαδή την επιρροή του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτή πρέπει να ενισχυθεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν η διαδικασία οδηγήσει μόνο στο να έχουμε ένα αδιαφανές παζάρι μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων δεν θα έχουμε καμία αξία στη διαδικασία. Για να υπάρχει πραγματική νομοποίηση πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και να τονίσω και την κοινωνική πτυχή. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα οποία αναφέρονται. Φτώχεια, ανεργία, κακές συνθήκες εργασίας, κοινωνικές διαφορές και εξασθενημένο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Όλα αυτά είναι πτυχές που έχουμε σκουπίσει κάτω από το χαλί παρά το ότι παίζουν τεράστιο ρόλο στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Το θέμα μας λοιπόν είναι εξίσου και η κοινωνική και η οικονομική κρίση. Και ένα σημαντικός λόγος γι' αυτό είναι πως οι κοινωνικοί εταίροι και οι εθελοντικές οργανώσεις στον τομέα τον κοινωνικό δεν έχουν σαφή ρόλο στη διαδικασία και αυτό το ρόλο πρέπει να αποκτήσουν. Χωρίς ενεργοποίηση στον τομέα τον κοινωνικό δεν θα έχουμε ποτέ ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κύριο Στόλογεν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την ε, κακή διαχείριση του οικονομικού ελλείμματος. Απλή απάντηση και τη δίνει η εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχουν πλέον ε, αυταπάτες ό,τι αφορά τα επιτόκια με τα οποία δανείζονταν τα κράτη-μέλη τώρα πλέον είναι επαρκές τα πιο κατάλληλα τα ε, επιτόκια. Επίσης έχουμε απαντήσεις μέσω της ε, προσπάθειας οικονομικής διακυβέρνησης, νέους κανονισμούς, νέες διατάξεις. Μεταξύ αυτών το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, που είναι και το βασικό εργαλείο για τη διαφορετική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος. Έχουμε και εμείς ε, ευθύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να καταστεί το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να επιμείνουμε επίσης και στην ευθύνη του Συμβουλίου, το οποίο πρέπει ε, δημοσία να δίνει λόγους επιχειρήματα για τα οποία έχουν ε, απορρίψει κάποιες από τις συστάσεις της Επιτροπής. Γκάλ Πέλτς τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Από τα σημαντικά έγγραφα για το Ευρωπαϊκό εξάμενο φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αλλάξουν ε, κάποιες επικεφαλίδες, κάποιους τίτλους ε, που έχει δώσει η Κομισιόν. Σήμερα η κρίση ε, αγγίζει τους πάντες, μικρά και μεγάλα κράτη και ίσως γι' αυτό γίνονται όλες αυτές τις προσπάθειες. Ε, τι δεν λειτουργεί τελικά, ιδέα όχι, είναι η εφαρμογή. Μίλησα και κατά το παρελθόν ε, για διάφορες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων. Έχουμε βουνά από χαρτιά μπροστά μας, αλλά αυτό είναι αυτό που θέλουμε τελικά. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μία αντιστοιχία και τα κράτη-μέλη δεν θα έπρεπε να εφαρμόζουν ε, μέτρα μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν άλλη ε, δυνατότητα, γιατί έχουν χρέος, ε, υπάρχει αυτή η επιβράδυνση της οικονομίας και θα πρέπει να δράσουν. Έχετε, ρωτώ την Κομισιόν, μία πρόταση. Πώς μπορεί να γίνει ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών, αλλά όχι σε ένα περιβάλλον στασιμότητας. Βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν συνενέσεις, θα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει προνομιακή θέση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο στα διάφορα θεσμικά όργανα και στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Στη διαδικασία Κατσδιάη το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γιασλοβιέσκα. Ευχαριστώ πολύ. Συζητάμε το οικονομικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τα μέσα τα οποία προτείνει η Κομισιόν είναι ένα ε, χρήσιμα, αλλά τελικά δεν αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Το ίδιο ισχύει από ό,τι αποδεικνύει η σημερινή συζήτηση και με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τις φωνές που ακούστηκαν εδώ και οι οποίες λένε ότι κάποια μέλη του Κοινοβουλίου συμμετέχουν ε, σε αυτές τις ε, συζητήσεις ενώ άλλα αποκλείονται από αυτές. Οι βουλευτές από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη ε, λέει ότι μπορεί να δημιουργήσουν διαιρέσεις και όχι τη, να βοηθήσουν την συνεννόηση στο κοινοβουλόγιο. στόχος είναι να βελτιώσουμε τα οικονομικά εργαλεία και αυτό είναι σκοπό και των χωρών μελών τη Ευρωζώνη και αυτών που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Και σίγουρα πρέπει να προασπίσουμε το κοινωνόμισμα. Ευχαριστώ. Κυρία Ζακονσάρη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στην ε, συνολική ενίσχυση της ε, ευρωπαϊκής ε, οικονομίας. Η μόνη αρνητική πτυχή είναι πως το κοινοβούλιο βασίζεται από ό,τι φαίνεται στο διαδίκτυο για ενημέρωση. Συμβούλιο και Κομισιόν μας λένε πως βιάζονται και υπάρχουν ε, τεχνικά προβλήματα. Μα αν είμαστε όλοι στο ίδιο τρένο θα πρέπει τουλάχιστον ε, να πηγαίνουμε και να ακολουθούμε τη σωστή γραμμή πέρα από την ταχύτητα του τρένου. Και όταν ορίζουμε την κατεύθυνση του τρένου, εάν προκύψει κάτι το νέο, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία του τρένου για να μην εκτροχιαστούμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φιγερέδο, ένα λεπτό επιμένω στο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε οι απαντήσεις του εκπροσώπου του Συμβουλίου για τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που στόχο έχει επαγρύπνηση, εποπτεία και παρέμβαση αντιδημοκρατική στις υποθέσεις των κρατών μελών για την κατάρτιση των εθνικών τους προϋπολογισμών δείχνει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι αυτής της πολιτικής διαδικασίας συγκέντρωσης των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών. Το τι συμβαίνει στην Πορτογαλία είναι ένα τρανό παράδειγμα για όλα αυτά. Μετά από... πρόκειται για μια τρομερή περικοπή κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων με περικοπές μισθών, βία μείωση του αγοραστικής δύναμη του πληθυσμού και των κοινωνικών παροχών. Αύξηση σε 2,5 ώρες εβδομαδιαίως ε, του ωραρίου εργασίας και γενική ε, φτώχεια του πληθυσμού ε, που τελικά συμβάλλει στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκανδαλώδης κατάσταση. Διακόπτη η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Φιγερέδο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σβάμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Συζητάμε την ε, στρατηγική του 2020, αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή. Εδώ πέρα μιλάμε για τεχνική οργάνωση και κύριε Ντομινίκ, έχετε δίκιο πως πράγματι δεν υπάρχουν κάποια μέσα για να ξεπεράσουμε την κρίση στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Μικρή μπορεί να είναι η συνεισφορά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για την κρίση κρίση. Οπότε θέλω να σα ρωτήσω, πιστεύετε ειλικρινά πω ο μακροοικονομικός διάλογο είναι κάτι το οποίο υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή. Πολύ αμφιβάλλω. Οι κυβερνήσει κάνουν προγράμματα για να επανεκλεγούν και δεν μπορεί να τι κατηγορήσει κανεί, Αλλά μακροοικονομικό διάλογο για τι μακροπρόθεσμε τάσει δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που πρέπει να το μάθουν ακόμα οι κυβερνήσεις. Δεύτερον, υποστηρίζεται άρα έναν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προπολογισμό για να εξισωθούν τα ελλείμματα στο επίπεδο των κρατών μελών και τρίτον υποστηρίζεται την απέτηση για μεγαλύτερη διακυβέρνηση της κοινή αγοράς με λιγότερους κανονισμούς και περισσότερη ελευθερία. Σας ευχαριστώ κύριο Σταμπάιντι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό που συζητάμε είναι σαν ένα άλογο που στην κτηνιατρική σχολή χρησιμοποιείται για να μελετηθούν όλες ε, οι αρρώσκες που μπορεί να έχει ένα ζώο. Αυτό το εξάμεινο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν επεύθυνες πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν μας δίνει αξιόπιστες πληροφορίες, δεν δίνει στο Κοινοβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά θα μπορούσε πιστεύω να καταλάβει η Κομισιόν ότι είμαστε σύμμαχοι, μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι της στην άσκηση του έλεγχου των κρατών μελών. Γι' αυτό χρειάζεται και ο δημοκρατικός έλεγχος. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας. Πρέπει να γίνει η κατάλυση έτσι και στα εθνικά κοινοβούλια. Κύριε Νταλή, τελικά τι συζητήσεις έχουν γίνει στα εθνικά κοινοβούλια για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύνοψη. Ματίας, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που φαίνεται από τη δήλωση του Συμβουλίου είναι ότι για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να θυσιαστεί η δημοκρατία όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό θέμα και η ερώτηση που θέτω είναι κατά πόσο θα υπάρξει συντονισμός πολιτικών χωρίς δημοκρατία. Πού είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πού είναι ο δημοκρατικός έλεγχος των Εθνικών Κοινοβουλίων για τις μεγάλες ε, ε, δημοσιονομικές υποθέσεις, αλλά μιλάμε για μια μεταβλητή τεχνική, γιατί γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο ελάφρυνε ε, πολύ τις συνθήκες για την, ε, στις χώρες που βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία όπως ε, η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ισπανία. Η Γερμανία έχει θέσεις για την Πορτογαλία αλλά δεν επιτρέπονται οι κρίσεις της Πορτογαλίας για την ε, Γερμανία. Και επίτροπε προσέξτε το αυτό. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα δημοκρατικής νομιμότητας ζητώντας από τους βουλευτές να πηγαίνουν να βρίσκουν τις πληροφορίες στο ίντερνετ. Εδώ είναι πρόβλημα. Είναι δημοκρατικός αποκλεισμός αυτό για το το οποίο συζητάμε. Τέλος του Κατσδιάη προσπάθησα να εξορροπήσω κάπως ε, τις ομιλητές από τις διάφορες ομάδες και δίνω το λόγο στον Επίτροπο Νταλή. Κύριε Νταλή, να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις παρακαλώ. Merci. Well, I would like to thank... Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση. Η ουσιοδέστερη αλλαγή που εισάγεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι το γεγονός ότι τώρα έχουμε Ευρωπαϊκό Συντονισμό των Φορολογικών και Δημοσιονομικών Πολιτικών πριν ε, ολοκληρωθούν οι εθνικές αποφάσεις. Μέχρι φέτος οι εθνικές πολιτικές, οι εθνικοί προϋπολογισμοί εκτιμώνταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού είχαν ληφθεί εθνικές αποφάσεις. Και αυτή είναι η μείζων αλλαγή. Αυτό το ανέφεραν πολλοί βουλευτές σήμερα, διότι αυτό ε, συνεπάγεται αυξημένη δημοκρατική ευθύνη για, τους, ε, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και βέβαια ε, σημαίνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικέ εθνικές συζητήσεις, ε, που είναι μια ανάγκη και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να την κάνουμε πράξη. Μέχρι στιγμή δεν θελήσαμε να αμφισβητήσουμε τις εθνικές πολιτικές στο δημόσιο διάλογο και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το Six Pack, οι δέσμε των έξι οδηγών, θα είναι σημαντικέ για να έχουμε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και για να μην δημιουργηθούν μακροοικονομικέ και δημοσιονομικέ ανισορροπίε σαν αυτέ που δημιούργησαν τη σημερινή κρίση. Έχετε δίκιο όμως. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων. Θα δώσει αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και την ανάπτυξη μέσα σε κάποια χρόνια. Ως εκ τούτου, πριν από δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε τον χάρτη πορείας για την σταθερότητα και την ανάπτυξη στοιχεία του χάρτη αυτού, του φύλου αυτού πορείας, θα παρουσιαστούν ε, και στην αυριανή σύνοδο ε, κορυφής. Φυσικά θέλουμε η Ελλάδα να επανέλθει στο μονοπάτι της ανάκαμψης, να δούμε τι θα γίνει με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και θέλουμε ε, τον τραπεζικό τομέα να τον ενισχύσουμε. Θέλουμε μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της οικονομικής διακυβέρνησης. Με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημειώνουμε ήδη πρόοδο για το τελευταίο στοιχείο. Δημιουργώντα μια πραγματική οικονομική ένωση. Εν τέλει, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαι πεπισμένο πω η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Το κοινοβούλιο σα έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στο να καταστεί πιο αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μεταξύ άλλων να ενισχυθεί και η νομοποίησή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν και στο μέλλον κρίσιμο σημαντικό ρόλο για να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση του συντονισμού των πολιτικών μας. Όλοι πλέον καλούμεθα να συνεισφέρουμε ώστε να πραγματοθεί αυτό ο σκοπό. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρο εκ μέρου του Συμβουλίου, ο κύριο Ντομινίκ. E, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και θέλω να ευχαριστήσω και όλους ε, τους βουλευτές που εξέφρασαν την αποψή τους για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το βασικό στοιχείο των περισσότερων τοποθετήσεων ήταν το δημοκρατικό στοιχείο της ε, διαδικασίας και το ποιος θα πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις. Συχνά έχω την ευχαρίστηση να συμμετέχω σε συζητήσεις ε, στο Εθνικό Κοινοβούλιο στην ε, Πολωνία και ακούω τα ίδια πράγματα κάπως διαφορετικά βέβαια. Τα Εθνικά Κοινοβούλια λένε πάντα πως θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στις ε, χώρες τους. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει στόχο ακριβώς αυτό όπως είπε ο Επίτροπος, ε, το Κοινοβούλιο έχει εμπλακεί πλήρως στην ε, διαδικασία αυτή και γνωρίζει τις απόψεις ε, των οικονομιών των κρατών μελών και γνωρίζουμε βεβαίως τις θέσεις των εθνικών κυβερνήσεων και υπάρχει βεβαίως κάποια αυτονομία εντός οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Γιατί το Εθνικό Κοινοβούλιο υιοθετεί τον Εθνικό Προϋπολογισμό και ο προϋπολογισμός είναι το βασικό μέσο οικονομικής πολιτικής. Οπότε δεν μπορώ να αποδεχτώ εγώ την άποψη πως δεν υπάρχει δημοκρατία γιατί βεβαίως αυτοί οι οποίοι ασκούν την μεγαλύτερη επιρροή στην ε, διαδικασία είναι τα εθνικά κοινοβούλια. Τώρα δεν ξέρω εάν μπορούμε να πούμε πως είναι μεγάλη ή μικρή επιτυχία το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Γιατί, γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν ξέρουμε πώς θα μεταφερθούν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εθνικό προπολογισμό των κρατών μελών όταν μιλάμε για μακροοικονομική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λοιπόν έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκει στη διαδικασία τα εθνικά κοινοβούλια και ε, τα εθνικά κοινοβούλια και τους άλλους εθνικούς φορείς ε, λήψης ε, αποφάσεων. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των ε, κρατών μελών και όπως είπε ο κύριος Επίτροπος ο έλεγχος ήταν ε, βεβαίως δευτερεύον αφού είχαν υιοθετηθεί όλα αυτά τα μέτρα Κομισιόν και Συμβουλίου δεν μπορούσαν να πούν πως τα μέτρα αυτά τα οποία είχαν ληφθεί ήταν ε, λανθασμένα, πως δεν θα ήταν θετικά τα αποτελέσματα Τώρα η διαδικασία έχει αλλάξει και τον τελευταίο λόγο έχει το πιο δημοκρατικό θεσμικό όργανο, δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία ξέρουν και καλύτερα το τι πρέπει να γίνει. Οπότε, κατά την άποψή μου, η δομή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η σωστή και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατηγορήσουμε τη διαδικασία αυτή για έλλειψη δημοκρατίας. Το πώς ε, θα εφαρμοστεί τώρα θα το δούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτού του σημείου και πηγαίνουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή την έκθεση του κυρίου Ριβελίνη για την απαλλαγή 2009. Και δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή κύριο Ριβελίνη. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.